τρομοκρατία ποτέ δεν έχει δικαιολόγηση και βρισκόμαστε στο πλευρό των Αμερικανών φίλων μας. Οι σκέψεις, ε, είναι, οι μας είναι κοντά τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωση του Πρωθυπουργού της Φινλανδίας κυρίου Γιούρκη Κατάινεν. Κύριε Κατάινεν, Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνοδεύει δε τον κύριο Κατάινεν και τον χαιρετίζω εδώ ο παλαιός φίλος και υπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Φιλανδίας πλέον, ο κύριος Αλεξάνδρ Στούπ. Πέσει στην έδρα του εδώ. και τον ρώτησα σήμερα πώς ξεκίνησε τη μέρα του γιατί ε, πάντοτε είχε μια σειρά στην, ε, στο Αστρασβούργο, εδώ, έκανε πάντοτε τη γυμναστική του και μου είπε ότι δεν την έκανε σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν. Δεν προβλέπεται διαδικασία λευκής κάρτας για τη συζήτηση. Χαίρομαι που έχουμε τον ε, κύριο Ζεμανουέλ Μπαρόσο επίσης, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον πρόεδρο. Το λόγο έχει. Όχι, ευχαρίστω. Αν θέλετε, χειροκροτήστε αν έχετε την ε, πρόθεση για τον κύριο Παρόσου. Ο κύριο Βέμπερ και ο κύριο Πέτερινγκ σημειώνω. Ε, άρχισε. και ο κύριο Κέλαμ. μα ξαφνιάζεται Θέλησατε να χειροκροτήσετε και εσεί. Κύριε Κάτάινεν, παρακαλώ, να λάβετε το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, όπως είπατε, ε, χτες είχαμε πολύ ε, σοκαριστικά νέα ε, σε αυτή τη βομβαρδιστική ενέργεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δύο τουλάχιστον πέθαναν και 140 τουλάχιστον τραυματίστηκαν. Τους σκεφτόμαστε. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα για το τι συνέβη. Θα δούμε τι θα μας πούν και τι θα ανακαλύψουν οι Αμερικανικές αρχές αλλά όποια και να είναι η αιτία αυτών των βομβιστικών ενεργειών θα υποστηρίξουμε τους Αμερικανούς ε, φίλους μας. Αγαπητά μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Σούλτς για την πρόσκληση αυτή ε, και θα ήθελα να τονίσω ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα διότι ήμουν δραστήριος ε, για ευρωπαϊκά ζητήματα κατά τη διάρκεια του ενηλίκου βίου μου. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ε, διαπίστωσα ότι η δική μου γενιά είχε μεγαλύτερες ευκαιρίες από τις προγενέστερες. Εγώ μπόρεσα να ολοκληρώσω τις, ε, τη φίτησή μου στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και ως φοιτητή Εράσμους μπόρεσα να ολοκληρώσω τη, τις σπουδέ μου σε ευρωπαϊκά ζητήματα. Αυτό μου άνοιξε τα μάτια γιατί ζούσαμε μια περίοδο μεγάλης αισιοδοξία. Η Φιλανδία είχε προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε ολοκληρωθεί σχεδόν η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Προετοιμαζόταν η επόμενη ε, διεύρυνση. Σήμερα ζούμε πολύ πιο δύσκολες και ε, προκλητικές ε, συνθήκες, δύσκολη καιρή. Ε, ζούμε στα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μέλλον της Ευρώπης και γι' αυτό χαίρομαι γιατί μου δίνετε ευκαιρία να μιλήσω σε εσά αλλά και να σας ακούσω. Το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επισκιάστηκε από την οικονομική κρίση οι άνθρωποι ανησυχούν για, την, για τις δουλειές τους, τις συντάξεις και το μέλλον των παιδιών τους. Καταλαβαίνουμε γιατί ανησυχούν και γιατί ε, έχουν, ε, αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση με ένα αρνητικό θυμικό. Κατανοώ αυτή την ε, απεσιοδοξία, αλλά με ανησυχεί παράλληλα όλοι αναγκαστήκαμε να ε, φτάσουμε σε δύσκολες επιλογές κατά την ε, ε, χρηματοπιστωτική αυτή κρίση. Συνεπώς, ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός επικράτησαν. Αυτή η στάση δυναμητίζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην Ευρώπη. Άρα είμαστε περισσότερο εσωστρεφείς παρά εξωστρεφείς. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στις ακραίες φωνές να τις ακραίες φωνές να επισκιάσουν την Ευρώπη τη στιγμή που θα πρέπει να έχουμε μία αξιόπιστη και πραγματιστική στάση προς τα εμπρός. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε αυτή τη στάση να δυναμητήσει και να δηλητηριάσει την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δεσπόσει ε, αυτού του φάσματος, αυτό το φάσμα. Πολύ εκτός Ευρώπης λένε ότι θα πρέπει να φτάσουμε στη, στις Ενωμένε Πολιτείε της Ευρώπης εδώ και τώρα. Δεν κατανοώ ε, εκείνους που μιλάν για διχασμό μεταξύ Βορρά και Νότου. Εάν διχαστούμε τότε χάνουμε την βάση κοινών αξιών και την δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια κοινή Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, είναι καθήκον μας και μέλημά μας να βρούμε λύσεις στις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις της Ευρώπης. Πρέπει να εξηγήσουμε στους ανθρώπους γιατί χρειάζεται μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και οι Ευρωπαίοι να θεωρήσουν ότι η ολοκλήρωση είναι δίκαιη. Δεν είναι εύκολο αυτό το καθήκον, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που αποτελεί ευεργέτημα για όλους. Χρειαζόμαστε πραγματική ολοκλήρωση. Κατανοώ ότι τα κράτη-μέλη και οι πληθυσμοί τους δεν βρίσκουν ότι η ζωή είναι δίκαιη αλλά μπορεί η Ευρώπη να είναι πιο δίκαιη στο μέλλον. Νομίζω ότι μπορεί. Δίκαιη ολοκλήρωση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται σε κοινέ αξίες και κανόνες που θα την χάνουν της εμπιστοσύνης όλων. Μεγαλύτερη ολοκλήρωση και δίκαιη ολοκλήρωση σημαίνει ότι ε, κρατάμε τάξη στα του οίκου μας. Θα πρέπει να βασιζόμαστε μέν στους δε, αλλά δεν, θα μπορούμε, να αναθέσουμε προς τα έξω τις ευθύνες μας. Δίκαιη ολοκλήρωση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί κατά τρόπο ώστε όλοι να νιώθουν ότι έχουν μία κοινή βάση. Πρόκειται για θέμα δημοκρατικής νομιμότητας και ε, λογοδοσίας, καθώς και ε, διάθεσης του ανήκειν. Ζητώ λοιπόν να λάβουμε αποφάσεις με βάση τους κοινού κανόνες και να ζήσουμε με αυτούς. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε κοινέ λύσεις έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη. Για να είμαι σαφής, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, αλλά και περισσότερη εθνική ευθύνη. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς βλέπω τη δίκαιη ολοκλήρωση έμπρακτα. Θα ασχοληθώ με τρία ζητήματα και θα τα δω υπό την οπτική γωνία της δίκαιης ε, ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να τηρήσουμε τους ε, κοινούς ε, κανόνες και αξίες, ευρωπαϊκές αξίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν χώρο ελευθέρου εμπορίου. Πρόκειται για κοινέ αρχές Επίσης δεν θα πρέπει να δυναμητήσουμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε τη διαφθορά και το, τη, τον, το κράτος δικαίου, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους. Αντιμετωπίσαμε και, τους αντιμετωπίσαμε και θεωρούμε ότι η ολοκλήρωση βασίζεται στη δημοκρατία. Θα πρέπει να ισχύσει το κράτος δικαίου. Καταλαβαίνουμε ότι εάν ε, δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε δεν θα έχουμε κοινούς κανόνες και την κοινοτική μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν να μην θεωρούν κίνδυνο τα κράτη-μέλη μια στεναρή Ευρώπη. Το κράτος δικαίου και οι κοινοί κανόνες και θεσμοί προστατεύουν την Ευρώπη. Δεύτερον, θα πρέπει να εξεύρουμε την ε, σωστή ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη. Αποτελεί την πεμπτουσία της. Η Φιλανδία θέλει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο. Δεχόμαστε ότι θα είμαστε μεγαλύτεροι εισφορείς στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό αποτελεί μέρος της αλληλεγγύης για τις χώρες που χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική αρρωγή. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω των ε, μέσων διαχείρισης της κρίσης, των άμεσων, της άμεσης δανειοδότησης και της ΕΚΤ. Ο καθένας προσπαθεί να ε, ανταποκριθεί στα δικά του καθήκοντα και παίρνουμε και πολιτικές αποφάσεις όταν πρέπει. Η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει όταν η Ευρώπη, ένα μέρος της Ευρώπης χρήζει ε, βοηθείας αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ανταποκριθούν στα, στις οικονομικές απαιτήσεις, διότι οι εθνικές κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για τις εθνικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, θα πρέπει να φτάσουμε σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση γιατί αυτό θα ευεργετήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Πολλοί Ευρωπαίοι βρίσκονται χωρίς εργασία, ιδιαίτερα οι νέοι. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανεργία, διότι ε, πολλοί βρίσκονται σε δινή θέση. Την προηγούμενη εβδομάδα επισκέφτηκα τη Λισαβόνα, όπου μίλησα με φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Μου έκανε μεγάλη σημασία το ταλέντο τους, αλλά παράλληλα είδα ότι ανησυχούν ιδιαίτερα για το μέλλον. Καταλαβαίνω πώς αισθάνονται. Θυμάμαι και τη δική μας ε, οικονομική κρίση κατά τη δεκαετία του 90. Το 20% των Φιλανδών ε, αντιμετώπισε την ανεργία. Είχαμε χάσει το 10% του ΑΕΠ μας σε πολύ λίγα χρόνια. Βρισκόμασταν στο χείλος της αφαιρεγγιότητας. Τότε ήμουν φοιτητή και εγώ ίδιος και θυμόμουν ότι ποτέ δεν θα αποκτούσα εργασία ή δεν θα είχα το δικό μου σπίτι. Κανείς μας δεν ήθελε να αποφοιτήσει διότι ήταν πιο ασφαλές να παραμείνει στο πανεπιστήμιο. Όταν θυμάμαι αυτά τα δεινά χρόνια, ε, τα ξαναζώ σαν να ήταν μία ασπρόμαυρη ταινία. Εν πάση περιπτώσει τα καταφέραμε και βγήκαμε από την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να είναι άμεσο μέλημά μας η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν υπάρχουν θαυματουργά μονοπάτια για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Αν υπήρχαν θα τα είχαμε ήδη χρησιμοποιήσει. Θα πρέπει να επιδοθούν έξι δις ευρώ για την καταπολέμηση της ανεργίας και χαίρομαι διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την, το Ταμείο ε, Εγγύησης για τους Νέους. Αυτό που έχει σημασία είναι να ανταποκριθούμε στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστική έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Θα πρέπει επίσης να ανταποκριθούμε στις νέες τεχνολογίες και στις βιομηχανίες βασιζόμαστε στις μεταρρυθμίσεις και στον ανοιχτό ορίζοντα. Θα πρέπει να εργαστούμε με τις αγορές, όχι εναντίον τους. Κύριε Πρόεδρε, λάβαμε βασικά μέτρα για να προβούμε στην ανασύσταση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης. Εσείς προωθήσατε τα έξι και τα δύο νομοθετήματα αντίστοιχα. Η ε, εφαρμογή αυτών των κανόνων σημαίνει επώδυνες εθνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν θα λειτουργήσουν εν μία νυχτή, αλλά θα αποτελέσουν όθηση μακροχρόνια. Εάν όλοι ακολουθήσουμε τους νέους κανόνες, τότε οι οικονομίες μας θα γίνουν όλο και πιο εύρωστες. Δεν πρόκειται για οικονομική θεωρία, πρόκειται για κοινή λογική. Κύριε Πρόεδρε, η εσωτερική αγορά και η προώθηση του εσωτερικού ελεύθερου εμπορίου είναι αυτονόητες αξίες καθημερινός βίος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει, αλλά όχι αρκετά. Κυκλοφορούν ελεύθερα τα εμπορεύματα στην Ευρώπη, αλλά όχι οι υπηρεσίες και γι' αυτό θα πρέπει να τεθεί και αυτό σε εφαρμογή κατά τρόπον αποτελεσματικό. Η εσωτερική αγορά, η ψηφιακή αγορά ιδιαίτερω προσφέρει νέε δυνατότητε και για δημιουργία θέσεων εργασία και για ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι η ευρωπαϊκή ανάπτυξη μπορεί να σημειώσει αύξηση κατά 500, η ιστορική οικονομία μπορεί να σημειώσει ανάπτυξη κατά τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ στα επόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραγνωρίσουμε τη σημασία του ψηφιακού εμπορίου που χρειάζεται βέβαια και λειτουργική εσωτερική αγορά. Εμείς αρχίσαμε ήδη τη δουλειά, άρχισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρώτο, αλλά δυστυχώς δεν ε, αρκούν αυτοί οι ρυθμοί εργασία. Χρειάζεται περισσότερη νομοθεσία, ευφυής νομοθεσία, η οποία να ε, προσελκύει τις δραστηριότητες κατά τρόπον ευφύ. Έχουμε το δυναμικό Έχουμε το καθήκον μάλλον να απελευθερώσουμε το, συναμικό, το σημαντικό δυναμικό του ε, εξωτερικού μας εμπορίου για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πραγματοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου ελεύθερων συναλλαγών ε, θα δημιουργήσει δύο εκατομμύρια θέσει εργασία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ανοίξουμε τι αγορέ και να δώσουμε σε ευρωπαϊκέ επιχειρήσει τι ευκαιρίε που έχουν ανάγκη στα γαλλικά. Πρέπει να απελευθερώσουμε το τεράστιο δυναμικό ελεύθερου εμπορίου για τη δημιουργία θέσεων εργασία, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, εκτιμήσει τις νέες δυνατότητες και πιστεύω ότι θα πρέπει να μην καταφύγουμε στον προστατευτισμό και στους φραγμούς η εκκίνηση του ελεύθερου εμπορίου και των, διαπραγματε... διαπραγματεύσεων για το ελεύθερο εμπόριο και τι επενδύσει με τι ΗΠΑ και την Ιαπωνία είναι μια πολύ καλή είδηση, καλύτερη στο τελευταίο διάστημα. Και αυτό λοιπόν α συνεχίσουμε τι προσπάθειε, στα αγγλικά τώρα, για να ε, διευκρινίσουμε και τα ε, σημεία των λεπτομεριών, χωρίς όμως να ε, να προσκρούμε στα, στις λεπτομέρειες. Πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση, να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και να μην χρειάζεται να παρεμβαίνουμε για να διασώζουμε υπερβολικά μεγάλες και υπό ε, κεφαλοποιημένες τράπεζες. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι βουλευτές, τρία τελικά σημεία. Καταρχάς χρειάζεται μια πραγματικά ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη. Η ενέργεια είναι ε, ζωτική για την οικονομία. Ο παγκόσμιο ανταγωνισμό στον τομέα τη ενέργεια οξύνεται διαρκώ και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει τη θέση τη μέσα σε αυτόν. Πρέπει να αποφύγουμε τι ε, ε, επιδοτήσεις, τι ενισχύσει που επιστρεβλώνουν την αγορά και να κάνουμε περισσότερε επενδύσει στι υποδομέ για την ενέργεια, να βρούμε τι εναλλακτικέ με χαμηλέ εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και να αποκαταστήσουμε το αποτέλεσμα του συστήματο ε, εμποριών εκπομπών που συζητήσατε και εσεί εχθέ. Δεύτερον, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα βήματα στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει περισσότερε ευθύνε για την ασφάλειά τη και ω εκ τούτου θα πρέπει να εργαζόμαστε πιο στενά μαζί. Χρειαζόμαστε πιο στενή συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε με τις ε, προκλήσεις σχετικές με την ασφάλεια, να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά ε, όρια, τους φραγμούς τους οικονομικούς και να εξασφαλίσουμε και για την ε, βιομηχανία ασφαλείας και άμυνας μια ευρύτερη εσωτερική αγορά. Αυτά τα περιμένω να τα συζητήσουμε το Δεκέμβριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για τη διεύρυνση Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή Προ τι χώρε τι ε, τις υποψήφιες εκείνες χώρες που αξίζουν να γίνουν μέλη τη. Κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, οι προσεχείς ευρωεκλογέ, ε, σε ένα χρόνο από εδώ, και, από και τώρα έχουν τεράστια σημασία, θα αποτελέσουν ε, μια δοκιμή στη δημοκρατική νομιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το δημοκρατικό τη αίρεσμα. Ποτέ δεν αντιμετώπισε τόσο σωματικές προκλήσει όσο σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε και μάλιστα η Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσ προσφέρει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στον Ευρωπαίο πολίτη σε μεγέθη που δεν έχει γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν η Επίρο μα. Θα συνεχίσει να το πράττει μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναδυθεί μέσα από την κρίση ισχυρότερη. Θα χρειαστεί χρόνο. Ο δρόμο δεν θα είναι εύκολο. Αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που μα ενώνουν και όχι σε αυτά που μα ε, χωρίζουν. Θα πρέπει να αναπτύξουμε την κοινή αμοιβαία εμπιστοσύνη χωρίς ε, την οποία δεν μπορούμε να είμαστε ισχυροί και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της δικαιοσύνης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση γιατί αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κατάινεν. Και τώρα εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Πρόεδρος Βαρόσο έχει το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμα μέλη, προτού να ξεκινήσω την ομιλία μου θα ήθελα να εκφράσω την ε, συμπάθειά μας και τη συλληπιτήρια στα θύματα και τους συγγενείς των, χθεσινών βομβιστικών Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κύριε Πρωθυπουργέ, ήθελα να σα πω ότι ήταν ευχάριστο που βρίσκεται στην ευχαριστώ που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μα ο, ο Πρωθυπουργό τη Φιλανδία. Να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για την πολύ σημαντική προσωπική συμβολή του στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Ο Κατάινεν έχει δείξει μια σημαντική δέσμευση προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατία και ο διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με λίγα λόγια, ο Φιλανδό Πρωθυπουργό και η χώρα του είναι υπέρ τη ευρωπαϊκή Ένωσης που καταρχήν αποτελεί μια κοινότητα αξιών, μια ένωση, ενότητα αξιών. Και αναφέρθηκε στον ε, κράτος δικαίου δεν έχει σημασία το οικονομικό μέγεθο, ε, η ιστορία και η πολιτισμός ε, κάθε χώρας, διότι έχουμε κοινέ αξίες και τις μοιραζόμαστε όπως και κοινά συμφέροντα. Έχουμε ε, έναν κοινό σεβασμό προς όλα τα κράτη-μέλη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Φιλανδία έχει καταδείξει ότι δεν μπορεί μόνο μια χώρα να προωθήσει την όλη Οικονομική Ένωση αλλά και η Φιλανδία είναι αποφασισμένη να προωθήσει διάφορα ζητήματα όπως τη ψηφιακή ατζέντα, την ενιαία αγορά και ούτω καθεξής θέματα που αφορούν και το, τα θέματα της ε, εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής άμυνας ε, είναι θέματα τα οποία συμμετέχει. Ο Πρωθυπουργό έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα ζητήματα και το ίδιο κάνει και η Κομισιόν ειδικά αυτή την περίοδο όταν οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να προωθηθούν. Γι' αυτό λοιπόν μέσω των προτάσεών μας θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ε, φόρα αποφυγή, φοροδιαφυγή που ανέρχεται σε ένα 3 ε, εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Με άλλα λόγια χάνουμε από αυτές τις φόρα αποφυγές και φοροδιαφυγές ε, ποσά τα οποία ανέρχονται σε έναν ετήσιο προϋπολογισμό μας κάτι το οποίο μας ε, δημιουργεί ένα τεράστιο ένα βάρος. Θα πρέπει να μετατρέψουμε την καλή βούληση σε πράξη. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί των προτάσεων της Κομισιόν για μια ισχυρή εντολή προκειμένου να διαπραγματευτούμε με την Ελβετία και, άλλους, ε, και άλλες γειτονικές χώρες για την καταπολέμηση των βατών του ΦΠΑ. Ε, θα πρέπει να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουμε σε κοινέ δράσεις και να εφαρμοστούν οι οδηγίες και οι κανονισμοί για την φορολογικού ε, φορολογικούς Νομίζω πως η Φιλανδία με τη στήριξή της αυτού του κλάδου θα ε, είναι πολύ, πολύ σημαντικός σύμμαχος. Πρόεδρε, Πρωθυπουργέ, αξιότιμα μέλη σε μια πρόσφατη ομιλία που έκανε στο βιβλίο σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, τόνισα την θέση της Φιλανδία ως ηγετική ε, ως χώρα που ηγείται σχετικά με το, το θέμα του δίκτυα ανταγωνιστικότητας. Βρίσκεται τρίτη στον κόσμο. Ανά την Ευρώπη, όπου να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την κρίση και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας παγκοσμίω, πρέπει να ε, ε, πάρουμε κάποια διδάγματα από την φιλανδική εμπειρία είναι σκληρά μαθήματα. Μετά από την τραπεζική κρίση τα δεκαετία του 1990 η Φιλανδία ε, αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες και πρόθεσε μεταρρυθμίσεις για την, ε, στον οικονομικό τομέα και ε, πρόθεσε την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τώρα αποδίδουν και η Φιλανδία δείχνει την αλληλεγγύη της ε, με τις ε, χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η κρίση στην Κύπρο μας έδειξε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα και είναι κάτι επίγον να ε, υλοποιηθούν και να υπερβληθούν. Υπάρχει μια τελική συμφωνία για τον μηχανισμό εποπτείας. Η Κομισιόν θα υποβάλει προτάσεις για έναν ε, μηχανισμό επίλυσης αυτών των κρίσεων τον Ιούνιο. Ε, το πιο σημαντικό μου δίδαγμα από όλα αυτά έγκυται στο ότι δεν θα πρέπει να ε, θεωρούμε ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει μία και έξω. Είναι μία καθημερινή προσπάθεια και σκληρή δουλειά που απαιτείται και η Φιλανδία το έχει αποδείξει. Κύριε Πρόεδρε, η Φιλανδία έχει ξεκινήσει ένα διάλογο με τους Ευρωπαίους εταίρους, συζητάει τις ιδέες, τις ανησυχίες και ενεργά συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για το ρόλο του που έχει προωθήσει αυτή την προσέγγιση και την στενή συνεργασία ε, αλλά και τη φιλία. Ευχαριστώ τη Φιλανδία για τη δέσμευσή της ε, απέναντι στην Ένωση και σε ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαρόσο και τώρα το λόγο έχει εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο Πρόεδρος κύριος Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Πρωθυπουργέ, θα συμφωνήσω και εγώ με τις δηλώσεις των προελισσάντων ως προς τις επιθέσεις στη Βοστόνη, τις βασικέ επιθέσεις. Εμείς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουμε τη βούληση και τη δύναμη να καταπολεμήσουμε την, θα το πω, τρομοκρατία αυτή. Μπορεί να μην ξέρω από πού προέρχεται, αλλά δεν έχει σημασία. Από όπου και να προέρχεται δεν είναι δυνατόν σε μια κοινωνία ελεύθερη, άνθρωποι αθώοι που δεν έβλεψαν κανέναν, που απλώς βγήκαν στον δρόμο για να αθληθούν, να χάνουν τη ζωή τους. Μόνο και μόνο γιατί θέλαν στο όνομα της ελευθερίας να εκφραστούν μέσω του αθλητισμού. Είναι απαράδεκτο, πρέπει να καταπολεμήσουμε, να πατάξουμε αυτή την τρομοκρατία. Κύριε Πρωθυπουργέ, σα άκουσα με πολύ προσοχή και δεν θα σα ξαφνιάσω να σα πω ότι ε, συμφωνώ μέσα σε πολλά σημεία. Θα ήθελα ωστόσο και πάνω απ' όλα να μοιραστώ μέσα σε κάποιε παρατηρήσει και να κάνω κάποιε ερωτήσει. Ω προ το νόημα τη Ευρώπη, καταρχά. Η Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο από ότι ένα απλό διάβημα οικονομική ή εγχείρημα οικονομική ολοκλήρωση. Το είπατε κι εσεί. Είναι πάνω απ' όλα κοινέ αξίε η Ευρώπη και πολύ σωστά το ειπατε κι εσει ειναι πανω απ ολα κοινε αξιε η ευρωπη και πολυ σωστα το η Ευρώπη χωρί αυτά σήμερα θα βρισκόταν σε ακόμη δυνατότερη κατάσταση. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα της Ισλανδίας όταν πτώχευσε. Δεν θέλω να υποτιμήσω τις δυσκολίες της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, αλλά χωρίς την Ευρώπη πού θα βρίσκονταν. Αγαπητέ Γερκή, πιστεύω όπως και εσείς ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ακρότητες, τους εξτρεμισμούς και ο καλύτερος τρόπος να το πράξουμε αυτό είναι να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας, να είμαστε υπεύθυνοι αλλά και αλληλέγγυοι και πρέπει να προχωρήσουμε προ περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν πρέπει να το φοβούμαστε αυτό, δεν πρέπει να φοβούμαστε να πούμε τη λέξη αυτή σε μια δύσκολη περίοδο κρίση όπου ο καθένα αναδιπλώνεται. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και με μια οικονομική και φορολογική εναρμόνιση που δεν είναι ε, προσβλητική φράση, είναι μια ανάγκη. Πρέπει να συζητήσουμε την διάρκεια του χρόνου εργασίας, τις εβδομάδες των αδειών, την, ηλικία τη συνταξιοδότησης. Όλα αυτά πρέπει να τα προωθήσουμε σε κοινέ βάσεις, γιατί έχει δημιουργήσει νέες πρόοδους στην ιστορική αγορά, αλλά εξαιτία των μεγάλων αποκλήσεων έχει φέρει και ε, πολλές αντίξωες συνέπειες. Και εγώ ως ε, επικεφαλής επιχείρησης γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί μιλάω, γιατί από την άλλη πλευρά του Ρήνου έχουμε <clears throat> έναν ανταγωνισμό από ε, έναν ανταγωνισμό σε σχέση με τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Από τα 60 εκατομμύρια της δικής μου, της δικής μου επιχείρησης έχω ε, μάλλον του κύκλου εργασιών τη μου επιχείρηση, έχω 1,5 εκατομμύριο επιβάρυνση κοινωνική σε κοινωνικέ εισφορέ ε, εργοδοτικέ, ενώ εάν μετακινούσα από το Στρασβούργο στο Κέλ την επιχείρησή μου, από την άλλη πλευρά του Ρήνου, δηλαδή δεν θα είχα αυτή την επιβάρυνση. Αυτό πρέπει να τα λέμε ξεκάθαρα. Και έχουν, έχουν κλείσει πολλέ επιχειρήσει και κυρίε και κύριοι στην Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη, το καθένα στη γωνιά του αυτή τη στιγμή, καλούνται ε, αυτόνομα είναι μόνο του δηλαδή αρμόδια το καθένα για να δώσουν απάντηση σε αυτήν την κρίση. Συμφωνώ με τον κύριο Πρωθυπουργό ότι χρειάζεται μια Ευρώπη δίκαιη λοιπόν, γιατί έχουμε και μεγάλη ανεργία στην Ευρώπη, όπω έχουμε όμω και πολλέ θέσει εργασία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν, βρει, δεν εντοπίζονται στο ίδιο σημείο αυτέ τι θέσει εργασία με την ανεργία. Γιατί λοιπόν να μην δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση στην ανεργία. Δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση ενεργεία και γι' αυτό δεν έχουμε ένα κοινό όραμα, αυτό το όραμα που θα μπορούσε να προσφέρει η Ευρώπη. Όσον αφορά την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την έρευνα, την πολιτική τη συνοχή, έχουμε πολλού τρόπου μόχλευση και δράση για να ενισχύσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων. Εάν δεν έχουμε ευρωπαϊκή έρευνα, Αγαπητέ Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόσο, δεν έχει νόημα να μοιράζουμε κονδύλια σε κάθε κράτο μέλο από ένα πρόγραμμα έρευνα το οποίο δεν είναι πραγματικά ευρωπαϊκό. Πρέπει να δείξουμε την παρουσία και να προχωρήσουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Η στάθμιση μεταξύ τη εργασία και τη αγορά εργασία, η καταπολέμηση τη ενεργεία των νέων και εδώ ευτυχώ έχουμε υποστηρίξει την εγγύηση για την νεολαία και χαίρομαι που η κυβέρνηση σα την υποστήριξη. Την υποστήριξη, αλλά κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο του Κοινοβουλίου, Κύρια Πρωθυπουργέ, όπω και εσεί θέλει μια ισχυρή Ευρώπη, ισχυρά κράτη, ισχυρή, οικονομία. Για να τα καταφέρουμε αυτά πρέπει να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνε που ισχύουν, τη διαφάνεια χρειάζεται, πρέπει όλοι προπολογισμοί να είναι ισοσκελισμένοι, πρέπει να περιοριστούν τα ελλείμματα, γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να ξοδεύουμε προ τώρα πόσα παράγουμε και σε αυτό πρέπει να πούμε πάλι την αλήθεια, για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη που απαιτείται για τι επενδύσει. Ερωτώ όμω και πάλι αυτό θα αρκέσει. Υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν πληγεί βαρύτατα από την κρίση με επιτόκια για το δανεισμό, που ο καλύτερο επιχειρηματία με το καλύτερο σχέδιο και όραμα δεν μπορεί να το υλοποιήσει στην, Ευρώπη, στην Ελλάδα που επισκέφθηκα. Ένα επιχειρηματία που ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο μου είπε, κύριε πρόεδρε, τι να κάνω, να επενδύσω όταν έχω επιτόκιο δανεισμού 10 και 12%. Και η απάντησή μου ήταν όχι, δεν μπορεί να επενδύσει όταν έχει τέτοιου είδου χαρτοφυλάκιο με επιτόκια 10 και 12%. Δηλαδή στη χώρα αυτή πλέον δεν μπορεί να δημιουργηθεί σε θέση εργασία. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να καταπολεμήσουμε και θα ήθελα για να καταπολεμηθεί η ενεργεία των νέων επισημάνω ότι πρέπει να αναζητήσουμε τα εξή κύριε Πρωθυπουργό και ξέρω ότι ίσω κάποιοι να αισθανθούν κατάπληξη και αποτροπιασμό αλλά θα ήθελα να περάσουμε στη συζήτηση για την αμοιβαιοποίηση του χρέου στην Ευρώπη. Ήρθε η ώρα πλέον γιατί το επιτόκιο του επενδυτή πρέπει να είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη το ίδιο. Δεν είπα να είναι ομοιόμορφο, αλλά κύριε Πρωθυπουργέ, εσεί, σα ερωτώ, έχετε κάποια άλλη λύση. Γιατί αν υπάρχει άλλη λύση, πολύ φως να ακούσουμε. Γιατί θα ήταν πολύ εύκολο να άρουμε έτσι μεγάλο μέρο του χρέου, να απελευθερώσουμε από αυτό το άχθο τον επιχειρηματία επενδυτή και να μειώσουμε το κόστο των επενδύσεων. Αυτή βέβαια αυτός ο καταμερισμός του χρέους θα σημαίνει ταυτόχρονα και καλύτερη διακυβέρνηση, θα σημαίνει α, συνειδητοποίηση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που, έχουν, που, συσχετίζονται με τα δάνεια, έτσι ώστε ο καθένας να λαμβάνει και τις δικές του ευθύνες μέσα σε αυτόν τον επιμερισμό. Ε, αυτό σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίε και κύριοι, και χρειάζεται και περισσότερη συνοχή, περισσότερη ολοκλήρωση ευρωπαϊκή, ενοποίηση δηλαδή, και γι' αυτό Κλείνοντας, αγαπητέ φίλε, πρέπει να κλείσω ίσως πρόωρα την ε, ομιλία μου κύριε Πρόεδρε, αλλά συγχωρήστε το πάθος με το οποίο μιλάω. Αναζητώ νέες θέσεις εργασίας για τον κόσμο μας ε, κύριε Πρόεδρε και δεν είχα και όλο το χρόνο της ομιλίας. Αυτό που θα πρέπει να επικρατήσει πάνω απ' όλα είναι κοινή λογική. Η ιστορία αυτά μας έχει διδάξει ότι όσο πιο καλά συνεργαζόμαστε, τόσο, όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο πιο καλά λειτουργεί η Ευρώπη, τόσο πιο πολύ μας προστατεύει η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, ε, Κύριε Ντόλαγκ, ακόμα και οι επισκέπτες σας χειροκρότησαν. Καταπληκτικό αυτό, αλλά θα πρέπει να τους επισημάνω, κυρίες και κύριοι επισκέπτε, ότι δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό μας να παρεμβαίνετε με ε, έκφραση των πολιτικών σας απόψεων από τα θεωρία των επισκεπτών. Αυτό μόνο βουλευτές μπορούν να το κάνουν. Αν και μπορώ να ε, δείξω κατανόηση για τους λόγους που σας όθησαν να χειροκροτήσετε. Τώρα, εκ μέρους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο πρόεδρος της ομάδας, κύριος Σφόμποντα. Κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα ξεκινώντα να υπογραμμίσω τα όσα είπε ο κύριο πρόεδρο του Κοινοβουλίου για τη Βοστόνη. Ε, βέβαια τα θέμα μα συλληπιτήρια ε, στου οικείου των θυμάτων πάνω απ' όλα. Κύριε Πρωθυπουργέ. Μιλήσαμε για δίκαιη ολοκλήρωση. Αυτή ήταν η κεφαλίδα και συμφωνώ. Γιατί θα πρέπει να δώσουμε μάχη γι' αυτό το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια καταστροφική κατάσταση με υψηλή ανεργία, με, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής κρίσης, όπως είπατε και εσείς. Πολλοί πολίτες δεν είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πολιτικής και ούτε καν υπέρ της Ευρώπης. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Μετά τις ανησυχίες λοιπόν των ε, πολιτών, με βάση τις ανησυχίες αυτές, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε χωρίς να βασιστούμε στο λαϊκισμό. Μιλήσατε για την κατάσταση της Φιλανδίας, κύριε Πρωθυπουργέ, λίγα χρόνια πριν. Τότε δεν υπήρχε Ευρωζώνη και η Φιλανδία δεν ανήκε σε αυτήν. Στην περίπτωση της Λετωνίας μιλήσαμε για μια κρίση που δεν είχε να κάνει με την Ευρωζώνη. Άρα θα πρέπει να υπάρχει άλλου είδους, είδους αλληλεγγύη και λύσει σε ευρωπαϊκή βάση. Ζούμε σε μια κατάσταση ύφεση. Κάτι το οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη πάντα ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι θα αλλάξουμε την αγορά εργασίας τη στιγμή που ε, μειώνονται οι κοινωνικές παροχές όπως είδαμε και στην περίπτωση της Πορτογαλίας το, στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι πολύ καλό το ότι παρευρεθήκατε στην Πορτογαλία, αλλά ε, ρωτήσατε τους πολίτες τι σκέφτονται για την Τρόικα και για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στη χώρα τους, ως προς τα πακέτα δηλαδή που προώθησε η Τρόικα για την Πορτογαλία. Και το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι κάτι τέτοιο ήταν αντισυνταγματικό. Μιλάμε λοιπόν για ουσιώδεις αλλαγές. Δίκαιη ολοκλήρωση σημαίνει ολοκλήρωση μεταξύ βορρά και νότου. Εγώ έχω βρεθεί στη Φιλανδία και προσπάθησα να έρθω σε επαφή με οργανισμούς, με φορείς. Η Φιλανδία έχει πολλά να μας δείξει δεν πρόκειται για τον μακροοικονομικό αλλά και για το μικροοικονομικό τομέα. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα εταιρικά πρότυπα για να συνδράμουμε και τον Νότο και να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου. Ας δούμε τη μακροοικονομική κατάσταση. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος Ρεν μας λένε ότι το επόμενο εξάμεινο θα είναι καλύτερο. Αυτό το ακούμε πολλές φορές ε, δεν είμαστε στο τέλος του τούνελ και δεν βλέπουμε κανένα φως. Ακούμε μόνο πολλαπλές υποσχέσεις και η Τρόικα δυσλειτουργεί. Δηλαδή υπάρχουν εσωτερικές διαμάχες για το ποιος είναι υπεύθυνος. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για αυτές τις πολιτικές και δεν μας αρέσουν πολλά από αυτά που κάνει ο κύριος Ρεν, αλλά αυτός είναι υπεύθυνο, όχι η Τρόικα, η ΕΚΤ ή οποιοδήποτε άλλος. Μιλάμε για την Επιτροπή η οποία φέρει την ευθύνη Ας την αναλάβει την ευθύνη λοιπόν και βεβαίως το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει. Αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε αυτή την τάση διότι οι πολίτες ανησυχούν από αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης και δραστηριότητας. Τέλος, ως προς το στοιχείο της ανάπτυξης χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη έτσι ώστε οι πολίτες να δεχτούν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά από ψυχολογικής άποψης είναι δύσκολο εάν υπάρχει ελπίδα. Να ξέρουμε δηλαδή ότι στο τέλος μεταρρύθμισης υπάρχουν ελπίδες. Πολλοί λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την ανάπτυξη. Είδαμε λοιπόν ότι έχουμε χάσει ένα τρεις ε, χάνουμε ένα τρεις ετησίως και αν ένα μέρος είχε εισπραχθεί φορολογικά τότε θα μπορούσαμε να αποπληρώσουμε το χρέος ή τουλάχιστον ένα μέρος του. Όταν έγιναν αυτές οι δημοσιοποιήσεις, ο κύριος ε, Κάμπρον είπε καιρός να αφυπνιστούμε και να μυρίσουμε το φρέσκο καφέ. Δεν θα πρέπει όμως να το βλέπουμε κατά αυτό το τρόπο πάντα. Και βλέπουμε ότι τρώγοντας ε, έρχεται η όρεξη. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις και να δούμε πού έγκυται το πρόβλημα. Δεν χρειαζόμαστε μόνο υποσχέσεις. Μιλάμε για δίκαιη ολοκλήρωση. Δεν είναι δίκαιο ότι πολλοί πλούσιοι αποστέλουν τα χρήματά τους στους φορολογικούς παραδείσους, ενώ άλλοι μένουν αποκλεισμένοι. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έναν εταιρικό φόρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για μία αντιμετώπιση η οποία θα έπρεπε να είναι τύπου είπα ε, το Λουξεμβούργο άλλαξε τη στάση του, θα αλλάξει τη στάση της και η Αυστρία ως προς την ε, παροχή στοιχείων και ο Επίτροπος σε μέτα μας είπε ότι θα πρέπει να έχουμε μια κοινή στρατηγική. Ελπίζω να το αντιμετωπίσετε και εσείς και να μας υποστηρίξετε ε, πλήρως έτσι ώστε και οι Υπουργοί Οικονομικών να κάνουν κάτι έμπρακτα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι φορολογικές διαφοροποίησεις. Δεν χρειαζόμαστε έναν ενιαίο φόρο, αλλά έναν φορολογικό χώρο. Πολλές εταιρείες της Πορτογαλίας πάνε στην Ολλανδία όχι για να επενδύσουν, αλλά για να εξοικονομήσουν στη φορολόγηση. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε από πλευράς εθνικής ευθύνης. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα χαιρόμαστε πάρα πολύ αν αλλάζετε γνώμη για το τέλος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, γιατί και αυτό ανήκει στη δίκαιη ενοποίηση της Ευρώπης. Γιατί δεν ε, συμφωνείτε με τις άλλες χώρες. Ελπίζω να σας πείσουμε πολύ σύντομα. Και τέλος, μάλιστα, οι πρωθυπουργοί της Ευρώπης ανέλαβαν την ευθύνη για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουν πολύ περισσότερο και ε, συμφέρον και δέσμευση και ελπίζω και ευθύνη και αίσθημα ευθύνης και η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική για τα φορολογικά και η κοινωνική δικαιοσύνη ψηλά ε, ε, στην ημερήσια διάταξη. Εάν γίνουν όλα αυτά, πραγματικά θα βοηθήσουμε για μια δίκαιη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Αλλά σας παρακαλώ σκεφτείτε ότι στην Ευρωζώνη δίκαιη ολοκλήρωση σημαίνει πολύ περισσότερη ολοκλήρωση. Από τότε που θα μπορούσε η Φιλανδία να λύνει μόνη της τα προβλήματά της. Ε, το φιλανδικό παράδειγμα μάλιστα, αλλά με διαφάνεια, με δικαιοσύνη στην Ευρωζώνη και αυτή θα είναι μια πάρα πολύ καλή όθηση ε, προς τα ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Φερχόφστατ εξ ονόματος της ομάδας του. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς κύριε Πρωθυπουργέ ε, να σας πω ε, ότι συμφωνώ και η ομάδα μου και εγώ με τα όσα είπατε ε, και εσείς και ο κύριος Βαρόσο για την επίθεση στη Βοστόνη. Επίσης σας ευχαριστώ και για την ομιλία σας, για την παρέμβασή σας. Γνωρίζω ότι είστε εμπειρογνώμων στην καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού και βεβαίως έχετε να αντιμετωπίσετε εσείς εκεί τους αληθινούς λεγόμενους Φιλανδούς και ας είμαστε ειλικρινεί όμως, είναι και μια καλή ευκαιρία να αναγνωρίσουμε ότι η συζήτηση μαζί σας δεν είναι πλέον ε, μόνο ένα φιλανδικό πρόβλημα. Ούτε καν ένα παραδοσιακό βρετανικό φαινόμενο, αυτός ο ευρωσκεπτικισμός που βλέπουμε να αναδύεται και να αυξάνεται. Ξέρουμε ότι προχθές μόλις δημιουργήθηκε πριν από λίγες μέρες ε, ένα κόμμα στη Γερμανία, η εναλλακτική λύση για τη Γερμανία, ευρωσκεπτικιστές, ένα κόμμα που θέλουν να βγει από το ευρώ η Γερμανία. Και για ε, μένα αυτό που ζητούν δεν ζητούν εναλλακτική λύση για τη Γερμανία. Αυτοκτονία για τη Γερμανία, μήπως να αλλάξουν όνομα στο κόμμα. Αυτό προτείνουν ε, και ουσιαστικά είναι και ανοησία και βλακεία για τη Γερμανία. Τι θα κάνουμε, δύο κύκλους στο ευρώ, βόρειο και νότιο ή θα γυρίσουμε στα παλιά εθνικά νομίσματα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που προτείνουν είναι διάλυση του ευρώ. Και νομίζω έχει έρθει η στιγμή και είναι πρόσφορο το έδαφος για να το υπογραμμίσουμε ότι αν υπάρχει μια χώρα που θα πρέπει να φοβάται ένα τέτοιο σενάριο, αν υπάρχει μια τέτοια χώρα στην Ευρώπη που θα πληγεί από ένα τέτοιο σενάριο, ε, αυτή νομίζω η Γερμανία. Και αυτό που προτείνουν τώρα τι είναι. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, κατά τη γνώμη μου, είναι τραγωδία. Ε, ε, όχι μόνο για την Ευρώπη, για τη Γερμανία την ίδια. Είναι ε, η διάλυση της γερμανικής εξαγωγικής μηχανής και μπορεί να είναι το τέρμα του γερμανικού θαύματος αυτό. Γιατί τα λέγω αυτά κύριε Πρόεδρε. Διότι έχω και αποδείξεις. Έχω μια μελέτη που έκανε η δεύτερη μεγαλύτερη Ολλανδική τράπεζα, ε, ING, ε, το υποκατάστημά τη στο Λονδίνο, δηλαδή στο City του Λονδίνου έχουν κάνει αυτή την έρευνα. Πού θα γινόταν καλύτερη ανάλυση αυτών των πραγμάτων. Και τι λέει αυτή η ανεξάρτητη ανάλυση που έγινε στο City του Λονδίνου. Ότι αν διαλυθεί το ευρώ θα διαλυθεί και η οικονομία στην Ευρώπη με πρώτο θύμα τη Γερμανία. Φυσικά. Και ποια άλλα στοιχεία περιλαμβάνει η μελέτη. Προτείνω να κάνετε 80 εκατομμύρια αντίγραφα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να το στείλετε σε κάθε Γερμανό πολίτη. Να τα πείτε αυτά, να τα συζητήσετε με την Επιτροπή Προπολογισμών, λέει ο Πρόεδρο. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι σαφέστατες οι επιπτώσει. Τι λέγει λοιπόν η μελέτη που έγινε στο City του Λονδίνου. Ότι θα υποτιμηθούν κατά 20% ε, κατά μέσο όρο τα νομίσματα των χωρών που εισάγουν από τη Γερμανία. Δηλαδή θα τους κλείσουν όλες οι εξαγωγικές αγορές. Επίσης, ένα νέο γερμανικό μάρκο ε, αμέσως θα χάσει, θα υποτιμηθεί κατά 20%, θα ε, διολυστήσει σε ισοτιμία ένα προς ένα με το δολάριο και θα αυξηθεί κατά πολύ το κόστος της εισαγωγής κυρίως ενέργειας. Τελευταία συμπεράσματα της ίδιας μελέτης ε, λέγουν ότι η διάλυση του ευρώ θα δημιουργήσει συρρήκνωση του ΑΕΠ της Γερμανίας κατά 10% περίπου μέσα σε μία διετία και μόνο το ξέρω ότι επαναλαμβάνομαι. Αυτό δεν είναι εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτό που είδαμε προχτές να ιδρύεται είναι αυτοκτονία για τη Γερμανία. Εφιάλτης για την Ευρώπη και όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Διότι σε τούτη εδώ τη μελέτη ένα από τα μεγάλα θύματα θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι θα χάσει 5% του ΕΠΤΟΥ από τη μια μέρα στην άλλη, εάν διαλυθεί το ευρώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και πρωθυπουργέ, δεν χρειαζόμαστε εναλλακτική για τη Γερμανία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι εναλλακτική για την Ευρώπη. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Πολιτική ένωση δηλαδή, ε, ουσιαστική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, ε, ένα Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικό και χαίρομαι πάρα πολύ ακούγοντας τον Ζωζεφ Ντόλ που μίλησε για μια ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Χρειαζόμαστε τραπεζική ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Καθάρισης των Τραπεζών. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, συμφωνούμε όλοι. Είτε θα γίνουμε ε, τα Ηνωμένα Έθνη της Ευρώπης ε, ε, μια χαλαρή συνομοσπονδία εθνών κρατών ή θα γίνουμε Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης. Τη δική μου επιλογή την ξέρω. Ελπίζω να είναι και δική σας αυτή για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει εξ ονόματος των Πρασίνων ο Πρόεδρος του ο κύριος Κονμπεντίτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Γκίφερ Χόφστατ. Πρωθυπουργέ, 3.700 φορές μιλήσατε για κανόνες. Σας αρέσουν οι κανόνες, το καταλάβαμε. Είπατε ότι εδράζεται η δημοκρατία στους κανόνες, μάλιστα. Σε μια κοινότητα όμως υπάρχει ένας κανόνας που ενίοτε έχει περισσότερη σημασία από τους λογιστικούς κανόνες. Ο κανόνας ελεγγύης είναι. Εξάλλου, η χώρα σας, η Φινλανδία, χαρακτηρίζεται από μια κοινωνική συνοχή, από μια εντυπωσιακή αλληλεγγύη. Όμως, όταν εσείς έρχεστε εισέρχεστε μάλλον στον ευρωπαϊκό χώρο αντιλαμβάνεστε με κρύο τρόπο ε, την αλληλεγγύη. Θα μου πείτε φυσιολογικό είναι Φιλανδός είμαι, εντάξει. Αλλά έχει και επιπτώσεις αυτό. Ορισμένες φορές έχουμε την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβάνεστε επακριβώς τα διαμείβοντα στην ε, Ευρώπη. Έχω την εντύπωση ότι μιλάτε σαν εκπρόσωπος ε, ε, της Νόκια εδώ. Καλά Νόκια έχετε, τι άλλο θα είχατε. Είστε πραγματικός Φινλανδός, Νόκια θα έχετε. Τέλος πάντων δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα, όχι αληθινός Φινλανδός, πραγματικός Φινλανδός είπα, έχει διαφορά. Λοιπόν, σήμερα ε, αλληλέγγυα Ευρώπη χωρίς πραγματικό προϋπολογισμό δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Μιλήσατε για την ευρωπαϊκή ευθύνη, για την ολοκλήρωση, την περιφερειακή ολοκλήρωση. Δίκιο έχετε. Έχουμε κρίση όμως και αν αυτή η συλλογική ευθύνη δεν είναι μια ευθύνη η οποία έχει ως έκφανση έναν πραγματικό προϋπολογισμό σε ευρωπαϊκό χώρο θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Εάν αύριο δεν θα καταφέρουμε ο ευρωπαϊκός αυτός προϋπολογισμός προϋπολογισμός να μην είναι μόνο οι εθνικές συνεισφορέ, αλλά ένας ε, προπολογισμό όπου ε, θα έχουμε ιδίου πόρου και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε δεν πάμε πουθενά. Είναι απλούστατο το μήνυμα που θέλω να περάσω. Ξέρετε η Μάργαρετ Θάτσερ ποια ήταν η μεγαλύτερη νίκη της. Ποια ήταν η μεγαλύτερη νίκη τη. 27 παιδιά. 27 εθνικές κυβερνήσεις ενώθηκαν και υπερασπίστηκαν την ίδια αρχή. Δώστε μου πίσω τα λεφτά. I want my money back. Να λοιπόν. Ε, αυτή είναι πραγματική ευρωπαϊκή άμυνα και με τις άλλες χώρες. Αυτά διαπραγματευτήκατε για τον ε, προϋπολογισμό. Ιτήθηκε η ευρωπαϊκή ιδέα, ιτήθηκε η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και ελπίζω οι συνάδελφοί μας εδώ να απορρίψουν αυτή την πρόταση, να δεχτούν αυτή την ευρωπαϊκή εκεί. Ξέρετε γιατί, διότι δοθήσει τη κρίση με το, ο προπολογισμό που μα δίνεται με μείωση των διαρθρωτικών 20% για την Ελλάδα, εφιέστατο. 25% για την Πορτογαλία. Μα είσαστε καταπληκτικός. Λοιπόν, αυτά που προτείνετε σημαίνουν ότι η βάση που έχουμε έχει εκλείψει. Ο Ζώσεφ Ντόλ από τους Πράσινους ε, μας είπε ε, ε, αν δεν καταφέρουμε να προτείνουμε κάτι ουσιαστικό για να γίνει λιγότερο επαχθές ε, το χρέος μπορούμε να αποδώσουμε την ευθύνη στην ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε όμως ποιος πληρώνει σήμερα οι φορολογούμενοι και το άχθος αυτής της κρίσης είναι τόσο βαρύ που για να το επομιστούμε χρειαζόμαστε κοινό ταμείο δημοσίου χρέους για να απαλύνουμε αυτό το άχθος. Εάν πληρώναμε 1% λιγότερο ε, ε, για την αποπληρωμή δημοσίου χρέου ε, θα μειώνεται κατά 20 εκατομμύρια το δημόσιο χρέο. Ε, δύο ποσοστιαίε μονάδε για την Ιταλία, μείωση για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέου σημαίνουν 20 εκατομμύρια λιγότερο δημόσιο χρέο. Χρειαζόμαστε κοινό ταμείο αποπληρωμή των δημοσίων χρεών, αλλιώ δεν πάμε πουθενά. Πρωθυπουργέ, όταν μιλάτε για του κανόνε, να έχετε κατά νου ότι έχει ύψιστη σημασία ένα κανόνα το να αφήνουμε τις χώρες ε, να πηγαίνουν ναι, ευθεία σε έναν τείχο δημιουργείται ε, ε, πολιτικές προϋποθέσεις που, δεν είναι, που δεν είναι βιώσιμες. Μόνο οι ακραίες δυνάμεις θα υπερισχύσουν αν ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπεντήτ εκ μέρου ε, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Το λόγο έχει ο Πρόεδρο ο κύριο Κάλαναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, επιτρέψτε μου να ε, συμφωνήσω κι εγώ με όλα αυτά που ελέγχθησαν μέχρι τώρα. Να στείλω κι εγώ τα συλληπιτήριά μου στους Αμερικανούς μας φίλους για τα τραγικά αυτά γεγονότα που έλαβαν εχθές χώρα στη Βοστόνη. Τώρα, τα στοιχεία και οι ειδήσει που προέκυψαν ήταν πολύ δυσάρεστα για την Μάργαρετ Θάτσο και φαντάζομαι θα απολαύσατε την ομιλία του κ. Κονμπεντήτη. Η κυρία Θάτσο πριν από 25 χρόνια καθόρισε μια, ε, ένα νέο δρόμο για την Ευρώπη στην περίφημη και γνωστή τη ομιλία. Και ρίχνοντα το βλέμμα προ τα πίσω, αυτό που εντυπωσιάζει είναι πόσο ταιριάζει η ομιλία τη αυτή στα σημερινά γεγονότα. Και επιτρέψτε μου να παραθέσω ένα απόσπασμα. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε τώρα είναι να λάβουμε αποφάσει για το τι πρέπει να γίνει. Να μην αφήσουμε να μα καταστρέψουν ουτοπικοί στόχη. Η ουτοπία ποτέ δεν επαληθεύεται και ε, θα ήταν και ωραίο αν προέκυπτε. Ακόμα και σήμερα πολλοί εστιάζουν την προσοχή του σε αφηρημένε ουτοπικέ έννοιε για το πώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Για αυτού μόνο περισσότερη Ευρώπη είναι η απάντηση. Ε, τέλος παράθεσης. Ε, κύριε Πρωθυπουργέ, με τη βοήθεια τη δική σα τη κυβέρνηση. το Συμβούλιο κατέληξε σε πιο ρεαλιστικό δρόμο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Για τη δική μου την ομάδα θα πρέπει να σας συγχαρούμε γι' αυτό. Ελπίζω μόνο να μπορέσετε να πείσετε κάποιους από τους συναδέλφους σας στο ΕΛΚ για τον δρόμο που θέλετε να ακολουθήσετε, γιατί μοιάζει μερικές φορές το ΕΛΚ να θέλει να δαπανίσει περισσότερα χρήματα από τους σοσιαλιστές. Πολλοί μιλάνε για μια τρελή πολιτική, για τον φόρο χρηματοψηφιστικών συναλλαγών και εσείς και σωστά το πράτετε. Λάβαμε λοιπόν ε, πίσω ένα δρόμο τότε με τον Τελόρ, με ανταγωνισμό, με ανοιχτή αγορά, πρωταθλήτρια και η κυρία Τάτσερ, εναρμόνιση και δυστυχώ υπερβολικού κανονισμού. Ο πρώην Προεπίτροπο κ. Φερχόγγεν από του σοσιαλιστέ είχε υπολογίσει ότι οι κανονισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοστίζουν στι επιχειρήσει 6 δι ευρώ, 4 φορέ δηλαδή το ΑΕΠ τη Φινλανδία. Και παρόλα αυτά όμω συνεχίζουμε να θεσπίζουμε όλο και περισσότερου κανόνε για την οικονομία. Δεν τα καταφέρνει αυτή πια να ανταποκριθεί και έχουμε πάνω από 6 εκατομμύρια ενέργου. Ο Άινστάιν είναι εκείνο που είπε ότι ο ορισμό του παράλογου είναι να επαναλαμβάνει κανεί συνεχώ το ίδιο πράγμα και κατά κάποιον τρόπο να περιμένει τα, να ακολουθηθεί ένα διαφορετικό δρόμο. Τώρα λοιπόν καλούμεθα να αποφασίσουμε. Η Ευρώπη είναι η επιτομή της ουτοπικής σκέψης. Δεν λάβουμε υπόψη μας τις οικονομικές συνέπειες αυτών που αποφασίσαμε. βεβαίω και η κρίση χρέου ήταν το έναυσμα, αλλά ε, φτιάξαμε παλάτια πάνω στην άμμο. Ζακ Ντελόρ είχε πει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την ευρωπαϊκή κυβέρνηση και αυτό νομίζω ήταν σαφές ακόμα και τότε. Ε, ακρεφνείς, ε, αναμφίβολα εγκρίνουν αυτό το δρόμο που ακολουθείτε και θα με ενδιέφερε να δούμε τι είπε όταν βρέθηκε εδώ. Το 2006 λοιπόν είχαμε τότε την Baby Thatcher που μίλησε εδώ, τον Βέλγο Πρωθυπουργό, τον κύριο Φερχόφστατ, διερωτώ με τι προέκυψε από αυτόν τότε ο κύριος Στούμπα ε, είπε ότι ε, δεν είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί φεντραλιστές, υπάρχουν καλυμμένοι φεντραλιστές, όχι όμως ε, ακρεφνείς φεντραλιστές. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα θα το έλεγε στη Φινλανδία. Αν λοιπόν οι εθνικοί ηγέτες ήταν πιο ειλικρινείς πριν από 50 χρόνια, σήμερα δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή την κατάσταση. Το τελικό κόστος αυτού του ουτοπικού εγχειρήματο θα είναι τεράστιο για πάρα πολλές χώρες και κυρίως για τη δική σας τη χώρα κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί γνωρίζουμε πόσο αντιλαϊκά είναι τα μέτρα μέτρα διάσωση. Όσον αφορά βέβαια τη γεωγραφική σα θέση, η θέση των Φιλανδών γίνεται κατανοητή. Αλλά οι Φινλανδοί θεωρούν ότι τα δικά του τα χρήματα των φορολογουμένων πρέπει να πάνε σε άλλε χώρε. Γνωρίζω από τι παρατηρήσει ε, τη ε, Φινλανδή ε, Υπουργού Οικονομικών ότι δεν αρέσει αυτό. Πολλοί ξέρουν τι κοστίζει η συμμετοχή στο ευρώ μακροπρόθεσμα και πρέπει δυστυχώ να λάβουμε δυσάρεστε αποφάσει. Η προσοχή μα όμω δεν στρέφεται ποτέ στι πραγματικέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε Ευρώπη που είναι να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε έναν διαφορετικό κόσμο. Ο πρώην Επίτροπος, ο κύριος Μπόλκενστάιν, που είναι στη δική σα οικογένεια, κύριε Φερχόφτσα, την προηγούμενη εβδομάδα είπε πολύ σωστά ότι το ευρώ αποδείχθηκε ένα χάπι, ένα ε, υπνοτικό χάπι το οποίο οδήγησε στην Ευρώπη στο να λαγοκοιμάται και να μην μπορεί να ανακάμψει στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Ε, ε, υπόθηκε κάτι εκτός μικροφώνου, είστε πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν να αναδιαρθρώσουμε τις οικονομίες μας, να περιορίσουμε το κράτος. Αυτή είναι η λύση που χρειαζόμαστε για την Ευρώπη. Αλλά αν μάθαμε κάτι από τη ζωή της Μάργαρετ Τάτσερ είναι ότι οι αλλαγές μπορούν να υπάρξουν μόνο αν είναι κανείς πρόθυμος να αγωνιστεί για αυτές. Υπάρχει λοιπόν πραγματική βούληση για αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να φτιάξει μια πιο ισχυρή Ευρώπη, να μεταρρυθμίσει τις πολιτικές της για τον 21ο αιώνα, να αποκεντρώσει πρέπει η Ευρώπη τη δύναμή της και η Μάργαρετ Τάτσερ νομίζω ότι δείχνει το σωστό δρόμο. Δεν πρέπει να παραλαμβάνουμε τα ίδια λάθη του παρελθόντος, γι' αυτό λοιπόν ας οδηγήσουμε την Ευρώπη σε μια νέα κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο λοιπόν τώρα έχει ο ε, Πρόεδρος της ομάδας του ΕΣΔ, ο κύριο Τέρο. Εξ ονόματος της ομάδας. Ευχαριστώ ε, πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό Κατάινεν και άμα σταματήσει ο συνάδελφο, μπορώ να συνεχίσω να μιλώ κι εγώ. Yeah. Ναι, κύριε Φερχόφστατ, εντάξει, θα ξέρουμε αυτά που λέτε. Ο κύριο ε, Τέρχο, ευχαριστώ. Θα αρχίσω και πάλι από την αρχή. Θα ήθελα, έλεγα, να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό Κατάινεν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην ομιλία του έκανε λόγο για μια δίκαιη ολοκλήρωση στην Ευρώπη. Εκεί μπορεί να δίστανται φυσικά οι απόψεις ως προς τον ορισμό της οι διαφορές στο εισόδημα είναι δικιά κατά την άποψή μου. Ε, υπάρχουν ε, μεγάλες δυσκολίες ε, στην εσωτερική πολιτική και στη Φιλανδία και δεν ξέρουμε πόσο δίκαιη είναι η αντιμετώπιση αυτή. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να μιλούμε πάντα με ειλικρίνεια και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούσαμε και τις δικές σας απόψεις. Μπορώ να κατανοήσω ε, τα όσα λέτε ε, στις μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς θα μεταφραστούν ε, στην πράξη για τους πολίτες και τι επιπτώσεις θα έχουν. Πολύ συχνά και η κυρία Μέρκελ εκφράζει την επιθυμία της να υπάρχει μεγαλύτερη ενοποίηση, ολοκλήρωση στην Ευρώπη και τελικά να γίνει η Ευρώπη ένα μεγάλο ομοσπονδιακό κράτος. Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις για το μέλλον. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα μπορούσατε δεχομένω να μας πείτε τι εννοείται ακριβώς όταν ομιλείτε για δίκαιη ε, ε, ολοκλήρωση στην Ευρώπη. Με τελικό στόχο απότερο ποιον ε, η δίκαιη ολοκλήρωση στην Ευρώπη θα είναι τελικά ένα ομοσπονδιακό κράτος. Βεβαίω θα πρέπει να ενισχύσουμε τις κοινέ ευθύνε. Αλλά ποια γραμμή θα ακολουθήσουμε, τη Βρετανική ή τη Γερμανική. Ο κύριος Γκούστευσον από την ΚΟΕ, παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα με τη σειρά μου να αποτίσω φόρο τιμή στα θύματα της επίθεσης στη Βοστόνη. Στη συνέχεια θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό Κατάινεν ε, στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω ότι η Σουηδία και η Φινλανδία είναι γειτονικέ χώρες, έχουμε την γεωγραφική εγκύτητα, αλλά και την οικονομική εγκύτητα. Έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις ε, με την ε, Φινλανδία και εγώ όλος ιδιαίτερος, διότι γεννήθηκα στη Φινλανδία και στη συνέχεια μετακόμισε η οικογένειά μου στη Σουηδία. Ε, υπάρχει ομοφωνία στην ngl σε σχέση με την ε, σφοδρή κριτική κατά της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμφέροντα των τραπεζών φαίνεται να επικρατούν και οι απλοί άνθρωποι έχουν να αντιμετωπίσουν περικοπές μισθών, μαζική ανεργία ε, και υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. 26 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι άνεργοι. Ένας στους τέσσερις σχεδόν είναι άνεργο. Στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία το 50% σχεδόν των νέων είναι άνεργοι ε, και αυτό αντιστοιχεί σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι βιώνουμε μια βαθύτατη κρίση σε πάρα πολλές χωρές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και στη Νότια Ευρώπη θυμίζει το σκηνικό το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου ορισμένε φορέ. Ο Ερυθρό Σταυρό θα έχει δυσχερέστατο έργο τα επόμενα χρονιά, συνεχίσουμε έτσι. Ε, βλέπουμε επίση τι γυναίκε που πλήττονται δι από αυτέ τι νεοφιλελεύθερες πολιτικέ, ε, διότι μειώνεται η συμμετοχή του στην αγορά εργασία ε, και καταβαραρθρώνεται η οικονομική τους ανεξαρτησία. Χρειαζόμαστε λοιπόν κρατεέ κοινωνικέ υποδομέ, όχι μόνο για τι γυναίκε γυναίκες αλλά και για τους ηλικιωμένους και αντί να κάνουμε όλα αυτά μετακυλίουμε την ευθύνη προς την οικογένεια. Περιμένουμε οι συγγενείς να φροντίσουν τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες. Ε, ένας από τους βασικούς στόχους ε, λέτε ότι είναι η μείωση της φτώχειας ε, και η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης στη Φιλανδία και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναρωτιέμαι Πώς ακριβώς μεριμνά η φιλανδική κυβέρνηση με τρόπο ώστε να μειώσει τις ε, ανισότητες ως προς τα εισοδήματα, γιατί αυτό είναι στοιχείο κλειδί και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας περάσω σε κάτι εντελώς ε, διαφορετικό. Στις προγραμματικές σας ε, δηλώσεις μας είπατε ότι είστε υπέρ της επιβολής φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Παρόλα αυτά δεν μας είπατε ότι θα συνασπιστείτε με τις υπόλοιπε 11 χώρες που το επιθυμούν. Πώς ακριβώς θα υλοποιήσετε το στόχο σας. Μας είπατε επίσης ε, στην ομιλία σας ότι χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Εγώ θα έλεγα όχι περισσότερη Ευρώπη, διαφορετική Ευρώπη χρειαζόμαστε. Σα ευχαριστούμε κύριε Γκούσταυσον, η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να μου επιτρέψετε να ε, εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και ε, τις καλύτερες ευχές μου προς τους ε, τραυματισμένους. Ποτέ δεν θα αποκτήσει το πάνω χέρι τρομοκρατία. Συζητάμε βέβαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να σας πω ότι θα προσπαθήσω να πω την άποψή μου μέσα σε ένα λεπτό. Πιέζομαι πάρα πολύ τι, ποια είναι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοιάζει με σοβιετική αυτοκρατορία, μοιάζει με ένα ε, μόρφωμα που αγνοεί τις απόψεις των πολιτών, ε, τα αποτελέσματα των ε, δημοψηφισμάτων και μετά ζητάει να γίνουν νέα δημοψηφίσματα. κλέβει τις καταθέσεις απλών ανθρώπων όπως συνέβη στην Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγνοεί ότι υπάρχει εισβολή στην Κύπρο και δύναμη κατοχής στο Βορρά. Ε, αυτό που συνέβη με το ε, βραβείο Ειρήνης ε, είναι και αυτό απαράδεκτο. Το μέλλον της Ευρώπης είναι ζωφερό. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραπέει. Γι' αυτό λοιπόν και επικρατούν απόψεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα αισθανθείτε τώρα σαν να είσαστε στη Φινλανδία, γιατί οι επόμενοι ομιλητές, οι τέσσερις ομιλητές που θα ακολουθήσουν, είναι Φινλανδοί, είναι δηλαδή σαν να βρίσκεστε στο ε, κοινοβούλιο της ε, Φινλανδίας και μόνο αυτό, αλλά θα είναι και τέσσερις κυρίες που θα λάβουν το λόγο η μία μετά την άλλη. Θα ξεκινήσει η κυρία Κόρολα. Κυρία Κόρολα, ξέρετε, πρέπει λιγάκι να σεβαστούμε το χρόνο, γι' αυτό θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να παραμείνετε στο χρόνο που έχει προβλεφθεί για εσάς. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Κατάινεν, ε, μιλήσατε για μια πραγματική, ρεαλιστική και δίκαιη ολοκλήρωση της Ευρώπης σε καιρούς κρίσης. Οι λαϊκιστές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης μιλούν με συνθήματα. Εμείς ε, επικεντρωνόμαστε ε, προς την ανάπτυξη για να φύγουμε από τη λιτότητα και να βρούμε σοβαρές λύσεις στα σοβαρά προβλήματα στην Κροατία, όπου συνεδρίασε το Προεδρείο του ΕΛΚ, ο κύριος Ντόλη είπε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πραγματική οικονομία, ε, στην ανάπτυξη για να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Συνεχίζω στα φινλανδικά. Θα ήθελα να σας πω, λοιπόν, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι ε, η κυρία Θάτσερ και η Αγγλία ζητούσαν ανέκαθεν τα λεφτά τους πίσω. Βεβαίω δεν θα πρέπει όλα τα χρήματα να ρέουν προς τις Βρυξέλλε. Όλοι θέλουν τα λεφτά τους πίσω, όλες οι χώρες. Αλλά με προστιθέμενη αξία, με κέρδος, με ωφέλη για τις χώρες μας. Όχι τα μετρητά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να τηρούμε τους κοινού κανόνες και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό υποστηρίζω τα όσα είπε Γύρκη Κατάινεν. Η εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς μπορεί να μην είναι πολύ ελκυστικό θέμα ή ενδιαφέρον για τους πολλούς, αλλά δείχνει ε, κάτι το οποίο ζουν ε, καθημερινά στα πορτοφόλια τους οι πολίτες, γιατί δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, θέσεις εργασίας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και την ψηφιακή αγορά που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο η Φιλανδία και θέλω να τη συγχαρώ γι' αυτό την πατρίδα μου. Η ανάπτυξη ε, της ψηφιακής ε, αγοράς και η ολοκλήρωσή της δεν είχε τους ρυθμούς ε, που επιθυμούσαμε και υπάρχουν χώρες μέλη που φέρουν γι' αυτό την ευθύνη. Αυτό τον καιρό είμαι σκιώδη συγγήτρια από την ομάδα μου για την οδηγία σχετικά με τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και του copyright και έχω μιλήσει με πολλούς ενδιαφερομένους και πρέπει να σας πω ότι αυτός ο κλάδος της οικονομίας, η δημιουργία ε, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλές θέσει εργασίας και θα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα των παρόχων ε, περιεχομένου στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ σημαντική και για την οικονομία μας, για την ψηφιακή οικονομία και χρειαζόμαστε η βελτίωση των συνθήκων ε, λειτουργίας των παρόχων αυτού του περιεχομένου στο διαδίκτυο. Και επίσης θα πρέπει να διατηρηθεί και η ε, πολυγλωσία και η πολιτισμική ποικιλομορφία. Και υποστηρίζω και τον Αλεξάνδερ Στούπ για τη μουσική βιομηχανία. Ο Πρόεδρος, παρακαλώ καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι εισέρχεστε στην αίθουσα, ε, παρακαλώ να καθίσετε και να συμμετέχετε στη συζήτηση. Και θα παρακαλούσα τους κλητήρες του Κοινοβουλίου να ε, ε, το επισημαίνουν αυτό στους συναδέλφους που δεν το ε, ακούν, γιατί συνεχίζει τη συζήτηση. Παρακαλώ. τους κλητήρες, να πηγαίνουν στους συναδέλφους που μπαίνουν στην αίθουσα και να τους λέγουν να λάβουν τις αισθούς και να συμμετέχουν στη συζήτηση, άλλως να παραμένουν εκτός του ημικύκλου. Ο κύριος Σβόμποτα με ρώτησε για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός Κατάινεν δεν απαντάει τώρα μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου γύρου μιλητών, διότι μας είπαν οι πολιτικές ομάδες ότι ε, πρέπει να είναι κοινή η συζήτηση. Τουλάχιστον έτσι με ενημέρωσαν οι υπηρεσίες κύριε Σπόποντα. Γνωρίζετε πόσο με συναρπάζει ε, ε, η συζήτηση και οι συνεδρίες με το, και το περιβάλλον του Γενικού Γραμματέα φαίνεται έτσι αποφάσισε. η κυρία Γιακονσάρη. Ο κύριος Στέρχου προσπάθησε να παίξει το χαρτί του ομοσπονδιακού κράτους. Αν ε, προβλεπόταν ε, μπλε κάρτα θα ρωτούσα ποιος είναι ο ρόλος του κυρίου Τέρχου και ποιος είναι ο ρόλος της ε, κοινοβουλευτικής του ομάδας και του κόμματος του στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Παζάρι το έχουμε κάνει εδώ. Εκφράζω το σεβασμό μου προς τον Πρωθυπουργό κατά διότι μπόρεσε να πυροδοτήσει μια επικοδομητική συζήτηση και στη Φινλανδία και εδώ στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι τη σήμερον ημέρα οι ευρωσκεπτικιστές ε, βρίσκονται στα φώτα της δημοσιότητας ε, και αμφισβητούνται βασικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελευθερία μετακίνηση, ε, κράτος δικαίου. Πιστεύουμε ότι ε, το ειδικό βάρος των ε, πολιτών ε, θα ασκηθεί μόνο μέσω του διαλόγου. Άρχισε αυτή η συζήτηση για τους φορολογικούς παραδείσους και σκεφτείτε ότι πριν από λίγα χρόνια θα φαινόταν αυτό αδύνατο. ανοίγουν το τραπεζικό απόρριτο η Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Είναι πρωτάκουστο. Είδατε τις δηλώσεις του κυρίου Κάμερον, παραδείγματος χάρη αρχίζει να επικρατεί αυτή η ιδέα περί ε, ίσης μεταχείρισης ε, στην φορολογία. Σημειώθηκε πρόοδος ε, λοιπόν στην τελευταία σύνοδο των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων ε, και επιχαίρουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο, όπως και ο κύριος Σβόμποντα και ο κύριος Γκούσταυσον, το εξής εφόσον τα γεγονότα καλούν για μεγαλύτερη διαφάνεια, μιλώντας για το τραπεζικό απόρριτο, παραδείγματο χάρη, ή για έναν ηθικό πολιτικό βίο, όπως στη Γαλλία. Θα μπορούσε ενδεχομένως ε, ο Πρωθυπουργό να, να θεωρήσει τη στάση του για το φόρο επιχρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ίση μεταχείριση για τις, ε, τους φορολογικούς παραδείσους και για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εκ μέρου λοιπόν της ε, ομάδας των Ελευθέρων θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό κύριο Κατάινεν για το γεγονός ότι ήρθε σήμερα εδώ. Οι Πρωθυπουργοί των κρατών ε, βεβαίως είναι πολύ σημαντικοί προσκεκλημένοι για μας. Ε, σίγουρα δεν συμφωνούμε όλοι στα θέματα που συζητάμε. Εγώ θα ήθελα να έχουμε πιο συγκεκριμένα οράματα, γιατί τα χρειαζόμαστε τα οράματα πριν από ένα χρόνο αποτελούσε αν θέλετε μακρινό όραμα το να ασχοληθεί κανείς με τους φορολογικούς παραδείσους. Σήμερα ε, το όνειρο αυτό μοιάζει κάπως να αποκτάει σάρκα και οστά αλλά για να υλοποιηθεί πλήρως ε, πρέπει να υπάρχει και η βούληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ο ανταγωνισμός σε φορολογικό επίπεδο και η φοροδιαφυγή των ε, κρατών στα κράτη-μέλη έχουν οδηγήσει σε απώλεια δισεκατομμυρίων εσόδων στα κράτη-μέλη. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ε, συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων. Τα κράτη-μέλη στηρίζουν την Τραπεζική Ένωση όπως επίσης και την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων. Βεβαίω το τελευταίο ε, δεν ε, είναι ψηλά στις προτεραιότητες, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Κύριε Πρωθυπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται πλέον με το μέλλον της, δηλαδή με το κατά πόσον θα είμαστε σε θέση να συστήσουμε ένα ομοσπονδιακό κράτος ε, κατά πόσο θα μπορέσουμε να άρουμε τις ε, διαρθρωτικές ε, ελλείψεις που υφίστανται αυτή τη στιγμή. <clears throat> Και από αυτού χρειαζόμαστε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα. Συνάδελφος Χάση, παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, αν έχετε την καλοσύνη να καθίσετε. κυρία Χάση. Ευχαριστώ πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι κυρίες και κύριοι. Η φοροδιαφυγή ε, στην Ευρώπη ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Πώς θα έχουμε ολοκλήρωση στην Ευρώπη ε, όταν είναι πιο εύκολη η διακίνηση των κεφαλαίων ε, χωρίς να κλείνουν τα παραθυράκια και η φορολογική παράδειση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. δεν θα πρέπει να πούμε σε ε, μία κούρσα μείωση της φορολογίας, σε ένα φορολογικό dumping, γιατί χρειαζόμαστε και για τα επόμενα έτη την απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ενδιαφέρεται για τον απλό πολίτη αλλά θα πρέπει να έχει και τα στοιχειώδη ε, έσοδα για ένα κοινωνικό κράτος. Γι' αυτό θα πρέπει η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η φορολογική παράδειση να παταχθούν. Λυπούμε πάρα πολύ ε, για τα όσα αποφάσισε τώρα να μπει σε μία κούρσα τέτοια η κυβέρνηση Φιλανδίας. Ο κ. Φοντάνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, στη συζήτηση κάποιοι είπαν, εκπλήσονται πάρα πολύ που αυξάνονται τα ε, λαϊκίστικα ε, κινήματα στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι η Ευρώπη έκανε κάποια λάθη γιατί τελείως δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. στη δική μου τη χώρα, λόγω των πολιτικών της Ευρώπης, βλέπουμε επιτιδευματίες να αυτοπυρπολούνται. Να, αυτή είναι η ευρωπαϊκή πολιτική. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει δρόμο στον εμπορικό τομέα, πρέπει να προστατέψουμε την παραγωγή μας. Δεν μπορούμε πλέον να δεχόμαστε τον παράνομο, αθέμητο ανταγωνισμό από άλλες χώρες. Στον τομέα του Σέγγεν υπάρχουν και προβλήματα ασφάλειας. Ε, το Σέγγεν λοιπόν πρέπει να τον αθωρήσουμε. Το ευρώ ως είναι τώρα δεν λειτουργεί, κυρίως για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Ε, και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ασχοληθεί λιγότερο με τις τράπεζες, περισσότερο με τις επιχειρήσεις, να ενισχύσει τις επενδύσεις. Και μία τελευταία μου ερώτηση αντί να δίνουμε ένα δις Ευρώπη στην Τουρκία για να μπει στην Ευρώπη, γιατί αυτό το δις δεν το δίνουμε στους άνεργους και στις επιχειρήσεις μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε, τώρα δεν μπορούμε πλέον να δεχθούμε άλλε ερωτήσει. Κύριε Βαν Λάρσεν, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εκ μέρου των μη γεγραμμένων, ο κύριο Μπρόν. Ευχαριστώ. Η δήλωση του Πρωθυπουργού εμ, στις 26 Μαρτίου, που ήταν η προηγούμενη παρέμβασή του, μιλούσε για την περιφερειακή ολοκλήρωση που υποτίθεται ότι βασίζεται σε κοινέ αξίε. Μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοκρατία χάρη στην ελευθερία έκφραση, αλλά τα κράτη-μέλη τη τι κάνουν, φυλακίζουν όλου όσου ασκούν αυτό το δικαίωμα. Τα δικαιώματα που ενθουσιασμού υπερασπίζονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο φιλελευθερισμός ε, και ε, κοινωνικοί φιλελεύθεροι όμως δεν υπάρχουν. Ε, η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι παγκόσμιο ζήτημα και θα μπορούσε να μας πει ο Πρωθυπουργός την ίδια ομιλία που θα έλεγε οπουδήποτε μάλιστα. Τι είπε καταφέραμε με την περιφερειακή ολοκλήρωση. Ήραμε τους φραγμούς ανάμεσα στους, στις περιοχές, επιμέρους περιοχές και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταφέραμε έτσι να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Ο Πρόεδρος Ζακόπ, τον ομιλητή, σας ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Γκάλ Πέλτς, μέλος του ΕΛΚ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας και για το γεγονός ότι υπενθυμίσατε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση, για τη βαθιά ολοκλήρωση. Θα πρέπει, ας πούμε, μεταξύ άλλων να έχουμε αξιοπιστία. Και επίσης συμφωνώ ότι για να υλοποιηθούν οι προτάσεις θα πρέπει να υπάρχει μια γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική με ένα γενικό σύστημα στην οποία, ε, στο οποίο θα εντάσσεται αυτή και για να δοθεί απάντηση στην κρίση ε, θα πρέπει να συνεχίζουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις σαφείς όμως. Αποφάσεις με πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα. Δυστυχώς οι ολιγορίες είναι πολλές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε φορά φέρνει περισσότερες προτάσεις, ιδέες προς εξέταση, αλλά χωλαίνει πάρα πολύ η ε, υλοποίησή τους και η πρακτική εφαρμογή σημαίνει όλο και περισσότερο φόρτο και άρθρος για τους πολίτες, για τα κράτη, οικονομική επιβάρυνση και τελικά ε, η ανεργία καλπάζει και μάλιστα η ανεργία των νέων. Χαίρομαι που τονίσατε τα προβλήματα των νέων, αλλά δυστυχώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν έχουν άμεσες ε, συνέπειες, ούτε τα επιθυμητά ε, απτά αποτελέσματα θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια θέματα ε, ή κάπως γενικά και θεωρητικά. Χρειάζεται ουσιαστική δουλειά για να απαντήσουμε στην κρίση, να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και τελικά να λύσουμε όλα τα καυτά ζητήματα που μας απασχολούν. Συμφωνώ ότι εκτός από την ολοκλήρωση στην Ευρώπη θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση δικαιοσύνη, κοινοί κανόνες που να ισχύουν ε, για όλους, που να έχουμε όλοι συναποφασίσει αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας και οι κανόνες αυτοί να ε, ανταποκρίνονται και στις αρχές και τις αξίες της Ένωσης. Αυτό μας χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάξας τώρα.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 ένα στους πέντε νέους είναι άνεργος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται να τελειώνει η κρίση σιγά σιγά, όμως όχι η ανεργία. 56% των νέων στην Ισπανία είναι άνεργοι. Επίσης, 45% του μισθού των ενηλίκων παίρνουν οι νέοι. Αυτό ισχύει στην Αθήνα, στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Είναι επισφαλής αυτές οι θέσεις εργασίας. Ζητούν ελεημοσύνη, Υποτίθεται για να έχουν δουλειά. Έχουν ε, πλέον ε, δημιουργήσει μια ξεχωριστή κοινωνική τάξη. Ε, η σε όλους της Ευρώπης ενωθείται. Είναι το σλόγγαν μας πλέον η εργατική τάξη ε, ε, χρειάζεται στέγη, τρόφιμα και ρούχα. Αυτό το κατάλαβαν ακόμα και τότε στη βιομηχανική επανάσταση. Ε, η λύση για την Ευρώπη έγινε στη λύση κατά του προβλήματος της ανεργίας των νέων. Από τους μία εγγεγραμμένους ο κύριος Στάτλε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ε, με αναστάτωσε πολύ η ομιλία σας. Ε, στην Ευρώπη έχουμε χρηματοπιστωτική κρίση, διαρθρωτική κρίση και ποια είναι η απαντησή σας. Περιορίζεται σε τρία θέματα να έχουμε ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας. Τώρα να δούμε αν αυτό μπορεί να λύσει την κρίση. Δεν το πιστεύω, είναι βέβαια απαραίτητο. Και μετά προτείνεται συγκεκριμένη αμυντική πολιτική. Μα πώς θα λέτε με την αμυντική πολιτική να λύσετε την κρίση, να αντιμετωπίσετε την κρίση και λέτε μετά ε, διεύρυνση. Μα δεν έχουμε ε, αφομοιώσει την τελευταία διεύνηση και προτείνεται άλλη. Ούτε μία πρόταση δεν καταθέσετε για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Αναφερθήκατε μόνο σε ουτοπικές ε, σκέψεις. Ε, εγώ ως Αυστριακός απορρίπτω πλήρως την αμυντική πολιτική γιατί δεν θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κρίση και μόνο αυτό δεν θα δώσει και θέσει εργασία στους άνεργους στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία. Με τη νέα σας πολιτική τίποτα δεν θα γίνει. Στη τελική ανάλυση στην Ευρώπη Ευρώπη με την αμυντική πολιτική, θα επαναφέρουμε την ανταγωνιστικότητα. Ε, άλλα πράγματα χρειαζόμαστε και για αυτέ τι τρελέ αμυντικέ πολιτικέ τι οποίε παρουσιάσετε εσεί σήμερα εδώ. Το λόγο έχει εκ μέρου του ΕΛΚ ο κύριος Μίτσελ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι αν θέλουμε να ξέρουμε πού πηγαίνουμε θα πρέπει να θυμηθούμε από πού ερχόμαστε. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημα. Ξέρω ένα νέο Λιθουανό ηλικία 30 ετών που δεν ξέρει τίποτα ε, για το τείχος του Βερολίνου. Ε, δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας. Μας έχει κατακυριεύσει η λιτότητα, αντί να μιλούμε για εδραίωση, για τη σταθερότητα. Αλλά πάνω απ' όλα αρνηθήκαμε και αποτύχαμε να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο. Δεν λέω φρούδες ελπίδες ε, ε, λέμε συνεχώς τι κάνουμε, αλλά δεν εξηγούμε γιατί το κάνουμε. Επί μεγάλο διάστημα ε, ο κόσμος δεν πίστευε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε όλες τις εξουσίες για να ελέγχει το νόμισμα, τελικά το απέδειξε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δώσει ελπίδα, για να δώσει ενάβσματα. Δεν χρειαζόμαστε μόνο σταθερότητα, χρειαζόμαστε και ε, νέα όθηση και κίνητρα και ενάβσματα. Εντάξει, σταθερότητα. 30 δεύτερα έχω πρόεδρε, μου δίνετε λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω ότι σε σχέση με την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου θα πρέπει να ε, αποφασίσουμε αν χρειάζεται μια γερμανική Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Αποφασίσαμε για το νόμισμα, βάλαμε τα θεμέλια, αλλά ε, τώρα χρειάζεται η ανακεφαλαίωση των τραπεζών και η τραπεζική εποπτεία και εδώ να σταματήσουν ε, οι ρυθμίσεις. Από εδώ και μπρος χρειαζόμαστε κίνητρα, ενάυσματα και ο φορέας για να γίνει αυτό θα μπορούσε να είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ήταν ε, πραγματική, πραγματιστική αισιοδοξία ε, που διαπνέει το μήνυμα που μας μεταφέρατε. Θέλετε μια Ευρώπη να βασίζεται σε κοινέ ε, αρχές και κοινέ αξίες. Όπως ο Αλεξάνδρ Στούπ, πρώην συνάδελφος, θα ακολουθήσω και εγώ την απαρίθμηση. Χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Πρώτον, διαφάνεια. Ε, λόγω της ε, φοροδιαφυγής χάνονται εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Χρειαζόμαστε λοιπόν αξιόπιστα δεδομένα. ουδάλλως ε, δεν θα ξέρουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Την, τον περασμένο μήνα ε, είδαμε ότι εκεί που νομίζαμε ότι είμαστε ασφαλείς βούλιαξε το κυπριακό πλοίο. Δεύτερον, αλληλεγγύη χρειαζόμαστε. Ε, είναι αμφίδρομη έννοια. Χρειάζεται εκατέρωθεν δέσμευση για να λειτουργήσει. Ε, η αλληλεγγύη σε καιρό κρίση ε, συνεπάγεται επιπρόσθετη δέσμευση για να διεξαχθούν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Και πάλι χρειαζόμαστε ενημέρωση για την πραγματικότητα, για την πραγματική κατάσταση. Έχουμε διαθέσιμα κονδύλια ή πρέπει να κάνουμε σοβαρές προσπάθειες μέσω μεταρρυθμίσεων να αποκτήσουμε επιπρόσθετα έσοδα. Πλησιάζουμε σε ε, σημείο καμπή διότι αυτοί που καταναλώνουν τα λεφτά ε, θα υπερβούν το αριθμό αυτούς που ε, παράγουν προσόδους. Για να έχουμε αυτά αποτελέσματα πρέπει να αλλάξει αυτή η αναλογία. Όπως είπε και η Μάργαρετ Θάτσερ, ε, χρειαζόμαστε αλλαγή, αλλά όχι από τους ε, πολιτικούς. χρειαζόμαστε αλλαγή στην κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ τώρα πραγματικά να καθίσετε στις θέσεις σας. Ε, και να ακούσετε τον Πρωθυπουργό κύριο Κατάινεν. Περίπου 50 συνάδελφοι ε, ε, αυτό τον καιρό κάνουν ξεχωριστούς κύκλους εργασίας, συνεδρίες πολιτικής ομάδας και άλλα πηγαδάκια και διμερείς επαφές. Τι εντύπωση θα αποκομίσουν οι θεατές στα θεωρία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούν να συζητούν ε, συνάδελφοι μεταξύ τους σε ιδιωτικές συνομιλίες. Είναι αναξιοπρεπές αυτό όταν μιλούν οι συνάδελφοί μας στην Ολομέλεια. Κοιτάξτε, ε, κανονικά απαγορεύεται να χειροκροτούν όσοι είναι στα θεωρία, αλλά παρόλα αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο λοιπόν έχει ο Πρωθυπουργός κ. Κατανίν. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, γιατί αυτή η διάσταση απόψεων μου υπενθυμίζει και τη διαφωνία απόψεων που υπάρχει και στη δική μας την κυβερνητική, στον κυβερνητικό συνασπισμό. Εκεί εκπροσωπούνται σχεδόν όλες οι απόψεις και εγώ καλούμε να συμβιβάζω τις απόψεις αυτές, να βρω έναν τρόπο για να προχωρήσουμε. Βέβαια, ένα είναι μόνο ο Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η διαφορά με εσά. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στη Μάργαρετ Θάτσερ. Μου άρεσαν πολύ ε, τα σχόλια από εσά που αφορούσαν την κυρία Θάτσερ. Η κυρία Θάτσερ είπε ότι τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό, πρέπει να τα κερδίσουμε. Αυτό λοιπόν είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε μαζί της, τουλάχιστον σε αυτό που είπε. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω και κάποια άλλα θέματα που αναφέρθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε κανόνες και στο κράτος δικαίου μια Ευρωπαϊκή Ένωση με αυστηρούς κανόνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, εκπροσωπείται η σκληρή γραμμή στην Ευρώπη. Κάθε άλλο. Εγώ πιστεύω ότι το κράτος δικαίου μια αυστηρή βάση κανόνων, το να ζει κανεί με τους κανόνες, αυτή είναι και η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Είναι δηλαδή σαν να έχει κανείς ε, μια ποδοσφαιρική ομάδα και να παίζει ποδόσφαιρο χωρίς να ισχύουν και για τις δύο ομάδες οι ίδιοι κανόνες. Μα δεν βγάζει νόημα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν οι αξίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει η Ευρώπη της Δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει να ζούμε με βάση κοινού κανόνες και πρέπει να σεβόμαστε το κράτος δικαίου. Αλλιώς δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Είμαστε απλά μια ομάδα που χρησιμοποιεί ευχάριστα λόγια αλλά δεν δεσμεύεται από τους ίδιους στόχους. Γι' αυτό λοιπόν το κράτος δικαίου και οι κανόνες είναι πολύ σημαντικοί κατά την άποψή μου. Κατά τα άλλα, πάρα πολλοί από εσάς ανησυχούν όπως και εμείς για το μέλλον της ε, ε, κοινωνίας της ευημερίας. Ανησυχούμε μήπως ε, τελικά η εξυγίανση των δημοσιονομικών ε, σημαίνει ουσιαστικές περικοπές ε, στο κράτος ευημερία. Αλλά θέλω να σας πω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί για να μπορούμε να κερδίζουμε αρκετά χρήματα για το κράτος πρόνοιας. Κατά τα άλλα, το κράτος πρόνοιας είναι το προαπαιτούμενο για να ισχύουν για όλους οι ίδιοι κανόνες. Η δική μου χώρα εξαρτάται πάρα πολύ από το εξωτερικό εμπόριο. το μισή περίπου των εισοδημάτων μας προέρχεται από το εξωτερικό εμπόριο. Και αυτό σημαίνει ότι για να έχουμε ένα γενναιόδωρο κράτος πρόνοιας πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί όχι μόνο στην Ευρώπη και στο Βορρά αλλά γενικότερα. Η ε, ευημερία σημαίνει ότι υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα που δεν μπορούν να προκύψουν μόνο από τους Φινλανδούς φορολογούμενους. Πρέπει να προσθεθούν και άλλα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Κάθε χρόνο προβαίνουμε σε μεταρρυθμίσεις γιατί είναι καθοριστική η ανταγωνιστικότητα για να ενισχυθεί η ευημερία, το κράτος πρόνοιας που θα προσφέρει σε όλους ίσες ευκαιρίε. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς λόγους γιατί ε, περικόψαμε τον προϋπολογισμό κατά 3 περίπου 100% του ΑΕΠ πέρυσι. Το κάναμε αυτό για να διαφυλάξουμε το κράτος πρόνοιας. Επίσης ε, μειώσαμε τους φόρου έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουμε πολύ καλή εκπαίδευση και σύστημα παιδείας στην Φιλανδία, πολύ καλές ε, εφευρέσεις, καινοτομία. Επενδύουμε στο κράτος πρόνοιας εδώ και χρόνια και θέλουμε τώρα να επωφεληθούμε από την ευημερία, από ε, την παιδεία. Η φορολογική πειθαρχία είναι ο καλύτερος φίλος του κράτους πρόνοιας. Αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι απλά κοινό νους. Και κάτι άλλο. Αρκετοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην αμοιβεοποίηση, την αποκαλούμενη του χρέους, τη συλλογική ανάληψη. Εγώ πιστεύω ότι ε, στα ευρωομόλογα είδαμε τα αποτελέσματα. Κατά τα πρώτα χρόνια ύπαρξης του ευρώ, όλες οι χώρες που είχαν υιοθετήσει το ευρώ αποκτούσαν το χρήμα με το ίδιο κόστος και αυτό είναι τμήμα του προβλήματος. Γνωρίζω ότι δίστανται οι απόψει από αυτού, αλλά θέλω να σας πω δεν είμαι σίγουρος ότι η συλλογική ανάληψη του χρέους αυτό θα αποτελούσε τη λύση για τα προβλήματά μας. Ε, κάθε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να συγχέουμε τις βραχυπρόθεσμες δυσκολίες με μακροπρόθεσμες λύσεις. Αν υπήρχαν ευρωμόλογα ή αν πρόκειται να εισαχθούν ευρωομόλογα που θα είναι κοινά, αυτό για μένα σημαίνει να δημιουργούμε μία ε, θρησκεία χωρίς να λάβουμε άνουμε υπόψη μας το διάβολο. Δυστυχώς παρεμβάσεις ε, που εμείς δεν ακούμε, λυπάμαι πάρα πολύ, ο Πρωθυπουργό απαντά, κοιτάξτε, σε αυτή την κατάσταση ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση από την αγορά. Υπάρχουν λοιπόν ε, πολλά πράγματα, ασκείται τεράστια πίεση αυτή τη στιγμή. Όμως αν επιτρέψουμε στις δυνάμεις αγοράς και τις ε, χρηματοπιστωτικές δυνάμεις να επαναλάβουν αυτό που έκαναν κατά το παρελθόν, κατά τα πρώτα χρόνια ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μακροπρόθεσμα δεν θα βοηθήσει. Επίσης, ε, να σας πω, στην οικονομία της αγοράς πρέπει κανείς να γνωρίζει σε ποια εταιρεία θα επενδύσει κανείς τα χρήματά του. Και βεβαίως και ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι και ποικίλουν αυτοί από χώρα σε χώρα και από εταιρεία σε εταιρεία. Γι' αυτό εγώ θα απέδιδα μεγαλύτερη σημασία στην ανταγωνιστικότητα που είναι ο καλύτερο τρόπο ε, για να κινητοποιηθεί η οικονομία, να εξυγιανθούν οι προεπολογισμοί, αυτό που προσπαθούν πολλέ χώρε αυτή τη στιγμή να κάνουν και πολύ σωστά και ήδη βλέπουμε κάποια αποτελέσματα και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Πήγα στην Πορτογαλία, ήρθα σε επαφή με πολίτε και αποκόμισα την εντύπωση πάρα πολλοί ε, πολίτε ε, ε, πρόκειται να υποστούν μεγάλες απώλειες. Ε, αυτή τη στιγμή οι δυσκολίες είναι τεράστιες για τους Πορτογάλους και τους Ιρλανδούς γιατί οι πολίτες ε, έχουν ήδη καταπιεί το πικρό χάπι, έχει πέσει ο πυρετός, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται ο πυρετός. Και αν δούμε τις αντιδράσεις της αγοράς, τα εξαγωγικά στοιχεία για την Πορτογαλία, βλέπουμε ήδη εκεί κάποια αποτελέσματα. Απλά πρέπει να δείξουμε υπομονή. Δεν ζητάω βέβαια την υπομονή από τον απλό πολίτη, γιατί αυτός υποφέρει σε καθημερινή βάση. Όμως ποια είναι η ελλακτική λύση αν οι χώρες αυτές πάψουν να εξηγαίνουν τους προπολογισμού τους θα υπήρχε κανείς να τους δανείσει χρήματα δεν νομίζω άρα δηλαδή πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες όμως οι χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρέπει και αυτές να ε, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν τα σωστά αποτελέσματα Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Κάλανεν. Κοιτάξτε, το ευρώ και η Ευρώπη είναι πολύ σημαντική. Αυξήθηκε η ανταγωνιστικότητα ε, κάθε μέρα, κάθε χρόνο αγωνιζόμαστε για να βελτιωθούμε. Επίσης έχει βελτιωθεί το εξωτερικό εμπόριο, έχει ενισχυθεί το κράτος πρόνοιας και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά που είπε ο κύριος Βερχόφστατ, συμφωνώ με την άποψή του για τη σημασία του ευρώ. Εγώ δεν νομίζω υπάρχει καν λόγος να κερδοσκοπεί κανείς ε, με το ευρώ. Ε, αυτό απλά επιδεινώνει την κατάσταση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλά. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά από κάποια χρόνια η Ευρωζώνη και γενικότερα η Ευρώπη θα είναι πολύ πιο ισχυρές από ό,τι ήταν κατά το παρελθόν. Κατόπιν, τέτοισαν κάποια ερωτήματα σχετικά με τον φεντεραλισμό. Εγώ προσπαθώ να μιλάω με αριθμούς, με στοιχεία δεν μιλάω γενικά έτσι γενικά για το φεντραλισμό. Όταν με ρωτάνε αν είμαι φεντραλιστή ή όχι, του λέω τι εννοείται το φεντραλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη Γερμανία, ή μήπω ε, το Ηνωμένου Βασιλείου. Για τι είδου ομοσπονδιοποίηση, τι είδου φεντραλισμό μιλάμε. Ε, σε παλαιότερε ομιλίε μου προσπάθησα να πω τι χρειάζεται να κάνουμε στην Ευρώπη έτσι ώστε η Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο ισχυρή, πιο ενωμένη αυτή τη συζήτηση λοιπόν ας την επικεντρώσουμε σε συγκεκριμένα θέματα. Τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε, πού μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ο φόρος χρηματοψηφιακών συναλλαγών κατανοώ το λόγο ύπαρξής του σε επίπεδο αρχής δεν έχω αντίρρηση αλλά αν μεταφερθεί, αν εφαρμοστεί αυτός ε, στη Φινλανδία χωρίς να ισχύει στη Σουηδία ή στην Εστονία καταλαβαίνετε θα έχουμε μεγάλες απώλειες και αυτό θα ζημιώσει την οικονομία μας και δεν το επιθυμώ. Η φοροδιαφυγή. Κατανοώ αυτά που κάνουν οι ευρωβουλευτές για να την αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούμε στη σημερινή οικονομία της αγοράς να επιτρέψουμε να συνεχίζονται αυτά που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό. Άρα δηλαδή και αυτό είναι ένα τμήμα του να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστικοί να βρεθούν λύσει για τη φοροδιαφυγή. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δραστηριοποιηθεί επί του θέματο αυτού, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί ανεξάρτητα με το τι δυνάμεις εκπροσωπούμε, Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς είμαστε υπέρ της ε, δίκαιης αγοράς του θεμητού ανταγωνισμού. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπηρετήσουμε τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ Κατάινεν. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ αυτή η συζήτηση και ερχόμαστε στις ψηφοφορίες. Που θα προεδρεύσει ο κύριος Βιντάλκο, άνδρας τον οποίο δεν βλέπω.